για ε, τρόφιμα που προέρχονται από τη φυσική οδό, δεν υπάρχει λόγο ε, να μην μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ε, λυπάμαι λοιπόν που το Συμβούλιο δεν είναι σήμερα εδώ. Ελπίζω πάντω ε, το θέμα να λυθεί ευνοϊκά. Σα ευχαριστούμε για την παρέμβασή σα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι μάλλον. Αύριο στι 12 η ώρα. Λοιπόν, το επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Κράμερ για τις βιομηχανικές εκπομπές, ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρήπανσης. Αναδιατύπωση. Νομίζω ότι ε, αλλά, ε, αλλάζει ο Επίτροπος. Ε, καλωσορίζουμε λοιπόν τον αρμόδιο Επίτροπο και αρχίζουμε τη συζήτηση στο θέμα αυτό με την παρέμβαση του κυρίου Κράμερ. Έχετε τέσσερα λεπτά τώρα και δύο στο τέλος της συζήτησης. Για να κλείσετε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Κράμερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύσκολη ώρα. Ήλπιζα να δω να κερδίζει η Ολλανδική ομάδα στον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, να μην ήταν κακό ιονός. Μου δείχνετε κι εσείς ότι συμφωνείτε κύριε Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνουμε σήμερα ένα νομοθετικό πακέτο, μια δέσμη μέτρων που συζητούμε εδώ και δύο χρόνια. Πράγμα το οποίο βέβαια οφείλεται όχι μόνο στα πολλά διαφιλονικούμενα ζητήματα, αλλά και ότι ε, παρενέβησαν εδώ μεταξύ ευρωεκλογέ και ότι χρειάστηκε να προσαρμόσουμε ορισμένα ζητήματα, ορισμένε προτάσει. Πάντω βλέπω στην κατάσταση που έχουμε φτάσει τώρα ότι μπορούμε να ψηφίσουμε μία συμβιβαστική λύση, μία μια σειρά προτάσεων τις οποίες μπορούμε να κάνουμε δεκτές, έστω και αν θέλαμε ενδεχομένω σε κάποια σημεία μια διαφορετική διατύπωση, κάποιες διαφορετικές λύσεις. Καταρχάς, θα αναφερθώ στις οικολογικές εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις των βιομηχανικών μονάδων, που θα είναι καλύτερες από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εισαγάγει μια ε, εξαίρεση με τις τροπολογίες μας και αυτό απευθύνεται ως παράκληση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξασφαλίσει την ε, σειρά εκείνη των διατάξεων που θα επιτρέπει την βέλτιστη δυνατή και ε, την χρήση της τεχνολογίας εχμής από τις βιομηχανίες μας, από τις πολυάριθμες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, βιομηχανικές μονάδες τα επόμενα χρόνια, το ταχύτερο δυνατό. Είναι βέβαια δαπανηρό κάτι τέτοιο. Ίσως τίθεται σε κίνδυνο με τον τρόπο αυτό η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ευρώπης και με δεδομένη την οικονομική κρίση. Και χωρίς να θέλω να σας μιλήσω για τα προσωπικά μου, προέρχομαι από την πρώην Ανατολική Γερμανία, λαϊκή δημοκρατία τη Γερμανία, η οποία κατέρευσε μεταξύ άλλων και γιατί έχασε το τρένο τη τεχνολογική εξέλιξη και γιατί δεν παρακολούθησε τις εξελίξεις τεχνολογία. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή από το οποίο εξαρτάται η ίδια η επιβίωση ενός κράτους. Άρα πρέπει και τη τεχνολογία να προλάβουμε και ταυτόχρονα να προσθέσουμε το περιβάλλον μας μειώνοντας τις ρηπογόνες εκπομπές. Αυτό είναι ο πρώτο στόχο που εξυπηρετούμε. Το δεύτερο κομμάτι τη οδηγία είναι αυτό που έχει να κάνει με τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης όπου προβλέπουμε για το 2020 ή 2023 ανάλογα την, τον προσδιορισμό συγκεκριμένων οριακών τιμών που θα πρέπει να τηρούν αυτές οι εγκαταστάσεις. θα πρέπει να αναλογιστούμε εν προκειμένου και σε συνεργασία βέβαια με το Συμβούλιο το κατά πόσον μπορούμε να έχουμε φιλόδοξες ε, τιμές που ορίζονται στην ομοθεσία, που βεβαίως θεωρούνται ευπρόσδεκτες και που βεβαίως όλοι υποστηρίζουμε κτλ. που όμως όταν έρχεται τη στιγμή να υλοποιηθούν, αποδεικνύονται εφιάλτης και ως προς το κόστος και ως προς το περίπλοκο της ε, ε προσαρμογής και ως προς τις αυστηρές κυρώσεις που επιβάλλονται. Και που με τον τρόπο αυτό πλήττεται πολλές φορές και η ίδια η βιομηχανία. Γι' αυτό λοιπόν για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και εδώ έχουμε να κάνουμε κυρίως με τα εργοστάσια ε, καύσης άνθρακα κυρίως ε, έχουμε να κάνουμε με τις εγκαταστάσεις της ύψης της αυτή τη στιγμή τεχνολογία, της βέλτιστης και πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Πρέπει να κλείσει λοιπόν αυτή η δέσμη μέτρων, πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό που είναι ε, η καλύτερη λύση, η πιο σύγχρονη λύση, η λύση η οποία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα για το μέλλον. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία αυτά δύο χρόνια. Με στήριξαν όλες οι μεγάλες ομάδες αυτές με τις επιλογές. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ συνάδελφε. Θα ήταν πολύ χειρότερα αν είχαμε αύριο την έκθεσή σας ασφαλώς, τουλάχιστον για σας και για μένα. Ο κύριος Ποτότσνικο, Επίτροπος, παρακαλώ τώρα για να, για να μιλήσει το θέμα αυτό. Mr. Chairman, honorable members of European Parliament, uh, Αγαπητοί βουλευτές, αγαπητέ εισηγητά, καλησπέρα σε όλους. Και εγώ είμαι φίλαθλος. Και συμφωνώ μαζί σας. Αλλά έχετε υπόψη ότι νίκησε πολύ άνετα, 3-1 η Ολλανδία. Νομίζω ότι η πρόταση παρόλα αυτά που συζητάμε σήμερα αξίζει την, παρουσία, την παρουσία μας εδώ. Ε, είμαστε στο κατόφλι μια συμφωνία για τι βιομηχανικέ εκπομπέ που θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει την βιομηχανική ρήπαση από μεγάλε εγκαταστάσει με βάση του ε, ε, περιβαλλοντικού στόχου. Παράλληλα, δίνει ευκαιρίε για οικολογική καινοτομία και μεθόδου βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή σε σημαντικού τομεί τη οικονομία μα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο εάν δεν γινόταν σκληρή δουλειά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Κράμερ, καθώς και την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε ε, στην πρόταση οδηγία για τι βιομηχανικέ εκπομπέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η οδηγία είναι σημαντικό τμήμα ε, για τον έλεγχο τη βιομηχανική ρήπανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θεωρούμε ότι σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπως, όπου η βιομηχανική ρήπανση είναι πάνω από το 80% των ε, ε, εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα, πάνω από το 40% της παραγωγής σκόνης και πάνω από το 30% της παραγωγής οξυδίων του αζότου. Επίσης, η εφαρμογή των τοπικών επιπέδων οδηγεί σε διαφορετική εφαρμογή των κανόνων. Γι' αυτό, λοιπόν, ε, είναι ανεπαρκή ε, η σημερινή κατάσταση, όχι μόνο ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο, αλλά γιατί στρεβλώνει επίση και τον ανταγωνισμό. Η ενδυνάμωση δύο από τις βασικές ε, αρχέ τη νομοθεσία, την εφαρμογή των καλύτερων, των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, καθώ και αναθεώρηση των οριακών τιμών εκπομπών σε μεγάλου τομεί, είναι απαραίτητη προπόθεση και είμαι ευτυχή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτή την άποψη μαζί μου. Ε, θα εξασφαλίσουμε επίσης ε, υγιείς ε, βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προστατεύουν την υγεία των πολιτών μας και πετυχαίνουν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και ταυτόχρονα έχουν και την ευκαιρία να τονώνουν την παραγωγή. Αυτή η συμφωνία είναι βασική για την κυριότητα του περιβάλλοντος και κατ' επανάληψη ε, στα πλαίσια της ε, διαδικασίας ε, συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, πιστεύαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία, αλλά τα καταφέραμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, δέχεται το πακέτο το συμβαστικό, είναι συμβιβασμό Χρειάζεται συμβιβασμό ε, για να φτάσουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Ενθαρρύνω λοιπόν το Κοινοβούλιο να δείξει την ίδια στάση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δεχτεί δηλαδή αυτό το συμβιβασμό. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν, η κυρία Γκαρντίνη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά. Κυρία Γκαρντίνη, το λόγο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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω ε, την ικανοποίησή μου ε, προς τον εισηγητή και να τον ευχαριστήσουμε γιατί πραγματικά ξέρουμε ότι καταλήξαμε σε ένα απρόσμενο όπως φαίνονταν μερικές φορές αποτέλεσμα. Ε, υπενθυμίζω ότι η οδηγία αυτή θεωρείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο ζήτημα στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ακούσαμε αυτά τα οποία μας είπε ο επίτροπο, Είναι προφανές σε όλους ότι βρισκόμαστε απέναντι σε ένα έργο περίπλοκο το οποίο απέτησε πολύ χρόνο αρκεί να σκεφτούμε ότι έχουμε μια οδηγία από το 1996 ε, και ε, ε, και αυτή τη στιγμή έχουμε την πέμπτη πιο σημαντική τροποποίηση τη οδηγία για τι βιομηχανικέ εκπομπέ. Ε, μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία μιλούν από μόνα του ε, και δείχνουν ε, τι ελλείψει και τα προβλήματα αυτή τη νομοθεσία. Νομοθεσία δύσκολη ω προ την εφαρμογή τη. υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε η διαδικασία παράβαση κατά εννέα κρατών μελών και πραγματικά μερικέ φορέ οι διατάξει δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Όλα αυτά λοιπόν ε, απέτησαν συμπληρωματικές προσπάθειες, ε, όλα, όλα τα όργανα ε, έκαναν υποχωρήσεις, όλες οι πολιτικές ομάδες, όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες ε, και πραγματικά βρεθήκαμε όλοι απέναντι σε ιδιαίτερα δύσκολες επιλογές. Πρέπει όμως να πω σήμερα και αυτό θέλω να πω με ιδιαίτερη πεποίθηση Κατά την άποψή μου, καταλήξαμε στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, προστασία του αγωνισμού, προστασία του περιβάλλοντο, ε, προστασία τη βιομηχανική πολιτική, προστασία τη απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγματι, από τη μια Έχουμε μία οδηγία που επιβάλλει ε, κοινέ υποχρεώσει σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και από την άλλη μία οδηγία που ε, ε, προβλέπει την απαραίτητη ευελιξία. Εύχομαι ειλικρινά τα αποτελέσματα να είναι αμέσω ορατά και η μείωση των, του άκου σε διοικητικό επίπεδο, προστασία του περιβάλλοντο και ενίσχυση τη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σα ευχαριστούμε κυρία Γκαρτίνη. Τώρα εξ ονόματο των σοσιαλιστών το λόγο έχει για τρία λεπτά η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κράμερ για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει και για τις προτάσεις του. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά αυτή για την οδηγία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πάνω από 50.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδων θέσεις εργασίας και πολύ σημαντικέ επιπτώσεις στο περιβάλλον μας. Η νομοθεσία λοιπόν, όσο και αν δεν είναι ε, τέλεια, αποτελεί τεράστια προόδο σε σχέση με τα όσα είχαμε μέχρι τώρα και αποτελεί τη σωστή επιλογή, το σωστό δρόμο, την κατεύθυνση προς την οποία θα θέλαμε να προχωρήσουμε. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην ε, επιτρέψουμε για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα ε, εξαιρέσεις, διατάξεις εξαιρέσεως και ως ε, προς τις εκπομπές ε, θείου και ως προς εκπομπές οξυδίων του αζότου και πιστεύω ότι αύριο στην ψηφοφορία θα πρέπει να ορίσουμε ε, όπου χρειάζονται εξαιρέσεις πολύ αυστηρούς κανόνες για την εφαρμογή τους. Καλό θα είναι λοιπόν ο κανονισμός να είναι σαφής και οι εξαιρέσει που θα εισαχθούν να μην είναι πρόσφορες σε καταστρατήγηση. Τα έγγραφα αναφορά βέλτιστες ε, τεχνικές, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές είναι το μέσον εκείνο που θα μας επιτρέψει την ανάπτυξη των προϋποθέσεων για την βέλτιστη δυνατή προστασία από τις πιο ρηπογόνες εγκαταστάσεις και την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της νομοθεσίας ταυτόχρονα θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τον, την έμεση στρέβλωση του ανταγωνισμού, δηλαδή την εξασφάλιση ενός ισόπεδου πεδίου ανταγωνισμού, ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού, για την προστασία του καταναλωτή, για την προστασία των θέσεων εργασίας μας ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε, εξ ονόματος τώρα των φιλελευθέρων, το λόγο έχει ο κύριος Ντέιβις για 1,5 λεπτό. Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ πάντα με τον κύριο Κράμερ όσον αφορά ε, ε, τα ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ε, ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει να επιβάλλεται. Αλλά όσον αφορά το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. γιατί πραγματικά μπόρεσε να επιχειρηματολογήσει ότι όσον αφορά αυτή την νομοθεσία ε, η Γερμανία την εφάρμοσε πιο αποτελεσματικό από ό,τι τα άλλα κρατημέλη συμπεριλαμβάνοντα και το δικό μου. Εθνικιστικό, αν θέλετε, το επιχείρημα αυτό. Αυτό θέτει τη Γερμανία σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλέ πτυχέ τη περιβαλλοντική νομοθεσία. Πρέπει να είναι ισότιμο το πεδίο. Η νομοθεσία που ε, εφαρμόζουμε θα πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ισότιμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να προστατευτεί το περιβάλλον και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, το γεγονό ότι ορισμένε χώρε δεν θα κερδίζουν ε, αγωνιστικό πλεονέκτημα με το να μην κάνουν συγκεκριμένε επενδύσει. Το ζήτημα είναι ότι τώρα εμεί προβαίνουμε στην αναδιατύπωση αυτή τη νομοθεσία δεν την χαλαρώνουμε, αλλά αντιμετωπίζουμε το γεγονό ότι τα πρώτα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη ε, βγήκαν από τη δύσκολη θέση. Το, ε, το, το, κράτος, το δικό μου κράτο μέλο, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έκανε αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει. Ρωτώ λοιπόν και θέλω να γραφεί στα πρακτικά. Τι περιέχεται σε αυτή τη νέα νομοθεσία που θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη στην ουσία θα πράξουν αυτό το οποίο πρέπει να πράξουν. Ευχαριστούμε κύριε Ντέιβις. Εξ ονόματος ε, της ομάδα των Πρασίνων, το λόγο έχει για 3,5 λεπτά ο κύριος Άικαουτ. Ehm, Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα εξαντλήσω τα τρία μου λεπτά γιατί εξακολουθεί να παίζει η Ολλανδία κατά της ε, Παραγουάης. Κερδίζουμε 3-1 προς το παρόν, άρα μάλλον έχουμε αγγίξει τον τελικό, αλλά παραμένει η αγωνία μας. Ήταν πολύ καλή λοιπόν η πρόταση αυτή που έχουμε να εξετάσουμε, ιδιαίτερα θετική για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, για την ποιότητα του περιβάλλοντος για τον καθένα και την καθεμία από εμά. Λυπούμε για τα όσα άκουσα από τον κύριο Ντέιβις, ο οποίος ε, λίγο πολύ ε, καταδικάζει την χώρα του, την κυβέρνησή του. Μπράβο κύριε Ντέιβις που τα είπατε τόσο ξεκάθαρα γιατί η κυβέρνηση σας είναι εκείνη η οποία ε, παρεμποδίζει την εξέλιξη στον τομέα αυτό. Έχουμε να κάνουμε τρεις ε, θερμοηλεκτρικές μονάδες που καίνε άνθρακα και που παράγουν περισσότερες ρηπογόνες εκπομπές από ότι όλες οι, θερμο, όλες οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες των κάτω χωρών μαζί. Πρέπει λοιπόν ε, να σφίξουμε λίγο τα λουριά και για τις μεγάλες βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι ναι μεν εμείς ε, στις κάτω χώρες ή τη Γερμανία έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία, ενώ αλλού στην Ιταλία, την Βρετανία είναι πολύ πιο χαλαρή η νομοθεσία. Πρέπει να σφίξουμε λοιπόν τα λουριά όπως έλεγα και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που πάντοτε ε, τραβάνε το χειρόφρονο στο Συμβούλιο για να παρεμποδίσουν τέτοιου είδου νομοθεσία, πρέπει πλέον να αλλάξουν στάση. Εγώ υποστηρίζω την μεταρρύθμιση. Ναι, προβλέπονται 12 χρόνια επιπλέον, αλλά όλες αυτές οι μονάδες που καίνε άνθρακα, είτε είναι στην Ιταλία, είτε στην Ινωμένη Βασίλειο ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, θα πρέπει πλέον να τηρήσουν χωρίς την παραμικρή παρέκκληση αυτού του κανόνε διότι έχει έρθει η στιγμή να τηρηθούν οι ίδιε διατάξει και οι ίδιε συνθήκε προστασία του περιβάλλοντο σε κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί οι πράσινοι βεβαίω υπερψηφίζουμε την νομοθεσία αυτή, όμω με βαριά καρδιά πρέπει να σα πω, διότι ακούμε διαρκώ να λέγεται ότι ε, πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των χωρών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να συζητήσουμε τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική, ο καθένας προσπαθεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της πατρίδας του. Και αυτό είναι λυπηρό. Είναι η στιγμή πλέον όλα τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές προστασία του περιβάλλοντος και αποτροπής της ατμοσφαιρικής ρήπανσης για να έχουμε καλό, καθαρό, καλή και καθαρή ατμόσφαιρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και ελπίζω και οι κάτω χώρες να πάνε στο τελικό και να κερδίσουν και εκεί. Ευχαριστώ κύριο Σκάλαναν για 1,5 λεπτό. Θα μιλήσω εξ ονόματο των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Ρεφορμιστών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω η απογοήτευση του κυρίου Άουκαουτ για την νομοθεσία που συζητάμε σήμερα το απόγευμα να μετριαστεί από αυτή την νίκη της Ολλανδίας που θα χρησιμοποιήσει ε, την, ε, τη βέλτιστη τεχνική. Δυστυχώς ε, η Αγγλία δεν προκλήθηκε, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Λοιπόν, όσον αφορά τη συζήτηση αυτή, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του δύσκολο το έργο, ε, δύσκολη νομοθεσία και προσπάθησε ε, να ε, λάβει υπόψη όλες τις απόψεις και κατέληξε σε κάτι το οποίο κατά την άποψή μου αποτελεί ένα αποδεκτό συμβασμό. Κανείς βεβαίως δεν, δεν κέρδισε απόλυτα. Ε, αυτό σημαίνει πάντα σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κανείς δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένος, ούτε τα κρατημέλη, ούτε και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Άικχαουτ είναι δυστυχής και αυτός. Ελπίζω αργότερα να ε, χαρεί με το αποτέλεσμα του αγώνα. Πάντως καταλήξαμε σε ένα συμβασμό που αποτελεί μια καλή ισορροπία κατά την άποψή μου. Από τη μια θέλουμε να προστατευτεί το περιβάλλον και από την άλλη να ληφθούν υπόψη ορισμένες ε, θεμητέ κατά την άποψή μου ανησυχίες ε, ορισμένων κρατών μελών για το γεγονός ότι ε, ε, εάν ε, κλείσουν εργοστάσια που χρησιμοποιούν άνθρακα, που καίνε άνθρακα και πάλι οι επιπτώσεις δεν θα είναι καλές, θα χαθούν θέσεις απασχόλησης θα, και θα υπάρξει πρόβλημα με τις εκπομπές. Και στην τελευταία ανάλυση μην ξεχνάμε ότι όλες οι βελτιώσεις που θέλουμε ε, όλε αυτέ τι βελτιώσει κάποιο θα τι πληρώσει. Στην τελευταία ανάγκη του καταναλωτέ έχουμε την ύφεση, άρα πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντο και ε, στι ε, δαπανηρέ βελτιώσει που απαιτούνται. Ευχαριστούμε ε, κύριε Κάλναν. Εξ ονόματο τώρα τη ε, Ενωτική Αριστερά, το λόγο για τρία λεπτά ο συνάδελφο Φεραίρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφε, κύριε Σιγητά, αυτή η νέα οδηγία θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πιο απαιτητικό σε ό,τι αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό βήμα για να υπεραπιστούμε καλύτερα το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υπεράσπιση των πληθυσμών που ζουν και δουλεύουν σε αυτές τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες ε, διαθέσιμες πρακτικές. Είναι σημαντικό να προσαρμοστούν οι μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες είναι πολύ ρηπογόνες ε, να σεβαστούν και να ενστερνιστούν αυτές τις βέλτιστες ε, διαθέσιμες τεχνικές. Είναι ένα μέτρο αυτό για να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις εγκαταστάσεις που έχουν πιο σημαντική επίπτωση, που είναι πολύ πιο σημαντικές θα πρέπει να δούμε την σημασία αυτών των τεχνικών για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση ρυθμιστική, κανονιστική, ε, που θα έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και που προστατεύει και την κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα ε, και στο περιβάλλον και στην υγεία και όχι τόσο σε μερκαντιλιστικές αντιλήψεις. Επίσης, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο ε, το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και τα αέρια που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές και να λάβουμε υπόψη μα όμω και τις διαφορές που υπάρχουν ε, μεταξύ κρατών μελών και να λάβουμε υπόψη και τι ιδιαιτερότητες των διαφόρων κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορετικέ ε, μέθοδοι παραγωγής. Υπάρχει επίσης διαφορετικό δυναμικό προσαρμογής και εστερνισμού των μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, αυτέ τι διαφορέ. Κάθε φορά στα εθνικά ε, μεταβατικά πλαίσια θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία για την εφαρμογή των ε, βέλτιστων ε, διαθέσιμων πρακτικών χωρίς να αμφισβητηθεί παρόλα αυτά η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επίσης θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μέτρα προστασίας πιο αυστηρά και θα πρέπει να εστιάσουν όπως είπα και προηγουμένως, και στα αέρια που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτά τα νέα ρυθμιστικά μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν εξυγχρονισμό των μέσων παραγωγής. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για τις πιο ευάλωτες οικονομίες. Θα πρέπει να εξασφαλίσω μια συνεχή βελτίωση της εφαρμογής των ε, βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών παντού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό ο κύριος Ρώση για να παρέμβει ο Ξενόματος Ευρώπης της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αυτή η νομοθεσία που εξετάζουμε σήμερα είναι ε, η πιο σημαντική νομοθεσία στη θητεία μα. Έχει σημαντικέ οικονομικέ επιπτώσει. Ξεκινώντα από ένα κείμενο το οποίο ψηφίστηκε στην Επιτροπή ε, με την αντίθετη γνώμη ε, τη αντιπροσωπεία τη Λέγκα του Βορρά, γιατί όπω προτείνονταν αρχικά θα οδηγούσε στο κλείσιμο πολλών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και στη μετατροπή άλλων μετά από την απόφαση του Συμβουλίου και στον τριμερή διάλογο ανάμεσα στην αρμόδια Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, αναθεωρήθηκε και τροποποιηθεί κατά την άποψή μα ε, με σαφώ ε, θετικό τρόπο. Σήμερα θα ψηφίσουμε ένα ε, κείμενο το οποίο ε, εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σήμερα διανύουμε μια περίοδο κρίσης. Όσον αφορά ε, το περιβάλλον και σεβασμός του περιβάλλοντος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουν ε, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί σε τελευταία ανάλυση θα μετατοπιστούν σε τρίτες χώρες, εκεί όπου δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί έλεγχοι. μάλιστα, η Κίνα πρόσφατα δήλωσε δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να μειώσει την, ε, το ποσοστό αυτό 80% άνθρακα, 20% πετρέλαιο. Αντίθετα, είπε ότι μέχρι το 2020 θα διπλασιάσει τις ενεργειακές ανάγκες. Το κλείσιμο λοιπόν ή η μετακατάσταση εργοστασίων ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμβάλλει στην ε, βελτίωση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, αντίθετα συμβάλλει στην επιδείνωση οικονομικής κρίσης. Ευχαριστούμε. τώρα θα προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις των συναδέλφων και πρώτα απ' όλα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σκύλα ο οποίος έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο και τον οποίο θα κληθούμε να υπερψηφίσουμε αύριο οριστικοποιεί το πλαίσιο για τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες. Αποτελεί μια νομοθετική επιτυχία γιατί σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών δυσκολιών αλλά και σημαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων προωθείται μια λύση λογική ρεαλιστική και ισορροπημένη. ιδιαίτερα αυτό ισχύει στην περίπτωση των εθνικών σχεδίων προσαρμογής που θα εφαρμοστούν στα μεγάλα θερμοελεκτρικά εργοστάσια. στη χώρα μου την ελλάδα οι αρχικές διατάξεις απαιτούσαν μια βίαιη προσαρμογή που, έθετε σε άμεσο κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ή εναλλακτικά θα οδηγούσαν σε εγκατάσταση νέων φίλτρων αξία εκατομμυρίων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα έμπαιναν σε παλιά εργοστάσια που θα έκλειναν σε τρία τέσσερα χρόνια. είτε δηλαδή θα είχαμε μια τεράστια σπατάλη ή ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. η αγορά κοινωνικο κοστο η αγορα ηλεκτρικου ρευματο δεν είναι δυστυχώ ακόμη ενιαία. θα χρειαστούμε καιρό για να φτάσουμε στο στόχο αυτό. αν λοιπόν επιδιώκουμε δρακόντιες ρυθμίσεις σε μία μόνο πτυχή της αγοράς τότε επιφέρουμε σοβαρό κόστος σε κράτη που είναι στην περιφέρεια της ένωσης και δεν έχουν ούτε τις διασυνδέσεις ούτε και την επαφή με την υπόλοιπη ενιαία αγορά. με το συμβιβασμό αντίθετα των εθνικών σχεδίων επιτυγχάνουμε έστω και με καθυστέρηση μεγάλα περιβαλλοντικά ωφέλη τα οποία επέρχονται σε διαφορετικό χρόνο με βάση τις πραγματικές περιστάσεις και συνθήκες που υφίστανται σε κάθε χώρα μέλος και χωρίς μεγάλο κοινωνικό κόστος είναι μια συνετή ρύθμιση για την οποία όσοι θερμά την υποστηρίξαμε έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι. ευχαριστώ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Έχει το λόγο ο κύριος Γιώλα Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Επίτροπος ε, Ποτότσνικ εξέφρασε ρητές ευχαριστίες προς το Κοινοβούλιο για την άτεγκτη στάση μας σε σχέση με αυτό το νομοθέτημα και για την ε, συμβολή που προσφέραμε για το μεγάλο αυτό άλμα προόδου για καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή κύριο Κράμερ, όλους τους και εισηγητές και όλους εκείνους οι οποίοι στήριξαν το στόχο του καθαρότερου ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. έχουμε δει και με τα οξύδια του θείου και με την σκόνη στον ατμοσφαιρικό αέρα ότι υπάρχουν μετρήσεις που δείχνουν ότι έχουμε αρκετά κακά επίπεδα, αρκετά δυσάρεστα επίπεδα ε, ρήπανση σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης. Τώρα έχει έρθει η ώρα, κύριε Επίτροπε, για σας, μετά την έγκριση της νομοθεσίας, να μείνετε άτεγκτος ως προς την υλοποίηση αυτής της νομοθεσίας, ως προς την παρακολούθηση της στήρησής της και οι πρόδρομες λεγόμενες ε, νομοθεσίες από τη δεκαετία του 90, 95 εδώ και 15 χρόνια που ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως γιατί ναι μεν μπορώ να δείξω κατανόηση ως προς τους Πολωνούς και τα άλλα νέα κράτη-μέλη αλλά τα παλαιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κανένα επιχείρημα για να δικαιολογήσουν την βραδιπορία τους ως προς την εισαγωγή αυτής της νομοθεσίας ό,τι και να λένε για θέσεις εργασίας και για οτιδήποτε άλλο δεν έχουν κάνει αυτό που έπρεπε να είχαν κάνει δεν έχουν φέρει εις πέρας το δικό τους καθήκον, που, καθήκον που ήταν υλοποίηση νομοθεσίας. Πολύ μεγάλη λοιπόν η επιτυχία. διότι έχουμε δει ότι πολλές φορές, δυστυχώς όπως συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, οι μεγάλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι απέφευγαν τις κυρώσει και τις υφίστανται μόνο οι μικροί, οι μικρότερες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος και τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να υπάρξει μείωση, επίεση ούτως ώστε να ε, μειωθούν ε, οι επικίνδυνες εκπομπές από τη βιομηχανία. Δεν πρέπει να περιοριστούμε σε απλώς ε, διοικητικά μέτρα και σε μια διοικητική προσέγγιση, γιατί μπορεί η υποπίεση να φτάσουμε σε μια δυσμενή κατάσταση μπορούμε να κλείσουμε κάποιες επιχειρήσεις, αλλά μπορεί μετά το κόστος ε, να είναι πολύ μεγαλύτερο όταν ψάχνουμε εκ των υστέρων να βρούμε την βέλτιστη λύση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούν και να ενστερνιστούν τις ε, βέλτιστες ε, τεχνολογίες και πρακτικές θα πρέπει όντω να βρούμε την καλύτερη λύση για να μειώσουμε τι εκπομπέ. Εγώ για 16 χρόνια ήμουνα ε, δήμαρχο και πρόεδρο μια περιοχή πολύ προβληματική ε, βιομηχανική και βρήκαμε κατόπιν δύσκολων συζητήσεων ε, φάνταστε λύσεις. Ευχαριστώ. Δύο λεφτά. Ο κύριος, η κυρία μάλλον, πιετικά είναι. Ευχαριστώ. Μιλάμε για τη σκόνη, ε, το θείο και τα οξύδια του αζότου. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις εκπομπές αυτές για, την για το ασφαλές περιβάλλον και την ασφαλή υγεία. στην Ευρώπη. Λυπάμαι που οι εξαιρέσει στο συμβιβασμό τελικά είναι πολύ μεγάλες. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τη βιομηχανία μας ή την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν νομίζω καθόλου. Αντίθετα. Στη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη, για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και την ανταγωνιστικότητα. Κάτι άλλο που με κάνει να λυπάμαι στην πρόταση αυτή είναι ότι δεν προοδεύουμε ούτε για το έδαφος, ε, ούτε για τις εκπομπές ε, που είναι επιβλαβείς για το έδαφος. Ελπίζω να προχωρήσουμε ε, με πιο γοργό ρυθμό για την οδηγία για το έδαφος. Παραδείγματος χάρη, όμως υπάρχει και ένα πράγμα που με κάνει να έχω κάποια αισιοδοξία. Το θέμα των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν αφαιθεί εκτός της οδηγίας αυτής, αλλά αυτή η οδηγία επιτρέπει παρόλα αυτά στα κράτη-μέλη να έχουν πιο αυστηρή νομοθεσία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Στο μέλλον, όταν, όταν θεωρηθεί αυτή η οδηγία, ελπίζω η Κομισιόν να εισαγάγει μέτρα για την εποπτεία των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Πάβελ Πόκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου προς τον κύριο Κράμερ για την ε, απίστευτη εργασία του ε, κυρίως σε διαπίπεδο διαπραγμάτευσης. Γιατί το να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό που χαρακτηρίζεται από τόσο μεγάλη ισορροπία, πραγματικά αυτό είναι υπεράνθρωπο έργο. Ε, η διατύπωση θα εναρμονίσει τις διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μειώσει το διοικητικό βάρος. Προφανώς ε, στη χώρα μου υπάρχουν ορισμένε πρωτοβουλίε των πολιτών, γιατί οι πολίτε μερικέ φορέ ε, ε, και σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένα δεν ικανοποιούνται ιδιαίτερα από το αποτέλεσμα του τριμερού διαλόγου. Ε, μπορεί βεβαίω να μην καταφέραμε τα πάντα, αλλά σίγουρα αυτό ο συμβασμό θα βελτιώσει το περιβάλλον και όχι μόνο στην Ευρώπη τα εθνικά σχέδια, τα μεταβατικά σχέδια θα επιβραδύνουν τη διαδικασία αυτή του συγχρονισμού. Αλλά ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα προσαρμογής στι οικονομίε που στηρίζονται στον άνθρακα. Επίσης, αποδυναμώθηκαν οι διεκδικήσεις όσον αφορά το δίχτυ ασφαλείας. Αλλά γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαναξιολογήσει τις ε, οριακές τιμέ και ε, άρα λοιπόν ε, θα καταλήξουμε τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα και πραγματικά ε, εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας κάποιος βαθμός ευελιξία. Μετά την αυρινή ψηφοφορία οι εθνικές αρχές θα αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Η αναδιατύπωση λοιπόν αυτή αποτελεί ένα ξεκίνημα, αλλά η πραγματική επιτυχία θα εξαρτηθεί από την συμμόρφωση και την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δύο λεπτά τώρα για τον κύριο Σόνικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. η εκπομπή βιομηχανικών καυσερίων πρέπει να περιοριστεί. Πρέπει να έχουμε πιο αυστηρές διατάξεις και εφαρμογή αυτών. Αυτό είναι ο κύριος στόχος τη νομοθεσία για τις βιομηχανικέ εγκαταστάσεις και τις εκπομπές ρηπογόνων ουσιών στην Ευρώπη. Η πρότασή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα συμβάλλει τα μάλλα στην βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια νομοθεσία η οποία θα καλύψει πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και όχι μόνο τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Ο τομέας της ενέργειας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καθώς δεν υπάρχει ενιαία ενεργειακή πολιτική υπάρχουν, επιβάλλονται διαφορετικές δια, τάξεις, αλλά πάνω απ' όλα εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα. Στην Πολωνία, Φερρυπίν, εξαρτώμεθα κατά ποσοστό άνω του 70% από την καύση του άνθρακα. Και μέχρι και 95% μάλιστα στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και με πιο ελαστικές διατάξεις και όρια για τις εκπομπές να μεταβούμε απρόσκοπτα σε ένα επίπεδο εκπομπών που θα είναι σύμφωνο με την νομοθεσία. Πρέπει δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, της κάθε περιοχής και η οικονομική τους ρόμη βεβαίως. Οι στόχοι που θα οριστούν θα πρέπει να είναι ε, δυνατόν να τηρηθούν από ένα κράτος μέλος χωρίς να δημιουργούν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Για ορισμένα κράτη-μέλη και λόγω της γεωγραφικής τους αλλά και λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δεν είναι εύκολο να τηρηθούν οι στόχοι. Ευχαριστούμε κύριε Σόνικ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Γκέρεκ komisja envi odrzuciła rozsądne mechanizmy dostosowawcze. przyjęcie η έκθεση Κράμερ θα θέσει τις ε, βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις σε μια δύσκολη θέση. Στην Πολωνία θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες ε, δυσκολίες ε, στο βιομηχανικό τομέα αν τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία από το 2016, πάνω από χίλιες εγκαταστάσεις στην Πολωνία θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως από οικονομική σκοπιά. Αυτός ο συμβιβασμός δημιουργεί μεγάλες ε, δυσκολίες, μεγάλες συγκρούσεις. Και θα μας ε, δημιουργήσει και τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας. Θα πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση αυτή γιατί δεν λαμβάνει υπόψη την εθνική μας πραγματικότητα είναι, κατα... είναι καθαρό ιδεολόγημα και δημιουργεί ε, στρέβλους του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ συνάδελφε. 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Σουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τελική συμφωνία ε, για την διατύπωση της οδηγίας όσον αφορά ε, τι βιομηχανικέ εκπομπέ είναι αποδεκτή και χαίρομαι ιδιαίτερα για την συμβαστική εργασία. Το τελικό σημείο περιέχει τα σημεία κλειδιά τα οποία υπερασπίστηκα και εγώ με του συναδέλφου μου στην ε, αρμόδια επιτροπή με στόχο το κείμενο αυτό να είναι φιλόδοξη νομοθεσία αλλά και ρεαλιστική. Πρώτα απ' όλα η διασφάλιση μια κάποια ευελιξία για τι επιχειρήσει και τι αρμόδιε αρχέ όσον αφορά την χορήγηση παρεκκλήσεων. Στη συνέχεια ήθελα να χαιρετήσω ε, την ε, νέα έκδοση η οποία είναι ιδιαίτερα, η ιδιαίτερα αλλά τώρα επιτρέπει να υπάρξει πολύ περισσότερος ρεαλισμός. Η συμφωνία επιτρέπει την καλύτερη σύνδεση ε, με την οδηγία για τις εκπομπές ε, και αποσύρει ε, από το κείμενο την, την λίγο σκόπιμη ιδέα της δημιουργίας μιας αγοράς ποσοστώσεων για τα οξύδια του θείου και του αζότου. Όμως, να μην ξεχνάμε τις διατάξεις που αφορούν το έδαφος. Η οδηγία για το έδαφος εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο αναμονής. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και δυστυχώς ε, θα πρέπει να, να το αντιμετωπίσουν μόνο τα κράτη-μέλη τα οποία ε, έχουν την κατάλληλη νομοθεσία, τη δική του νομοθεσία. Αύριο το Κοινοβούλιο ε, θα ψηφίσει τα στοιχεία στα οποία υπήρξε συμφωνία μετά από τον τριμερή διάλογο. Τεράστια εργασία όπου όλοι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να μην περάσουμε στη διαδικασία συνδιαλλαγή. Υπενθυμίζω, το κείμενο είναι κρίσιμη σημασία και για τη βιομηχανία αλλά και για την περιβαλλοντική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Σουλή. Και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η οδηγία για τη μείωση των ε, βιομηχανικών εκπομπών θα επηρεάσει διάφορους βιομηχανικούς τομείς οι εγκαταστάσεις ε, που καλύπτονται από την οδηγία θα πρέπει να λαμβάνουν μία άδεια ε, για τις οριακές ε, τιμές εκπομπών και θα πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Για να λάβουν αυτές τις άδειε, οι εταιρείε που καλύπτονται από την οδηγία θα πρέπει να έχουν σχέδια εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, κάνοντας τις κατάλληλες επενδύσεις για να μειώσουν τις εκπομπές. Αυτή, αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να συμπληρωθεί και από μια βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία, ούτω ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, αλλά διατηρώντας τη βιομηχανική της παραγωγή και διατηρώντας και το εργατικό της δυναμικό εδώ, ταυτόχρονα με τη μείωση της μόλυνσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη σε πολύ πρόωρη φάση για να ρυθμιστούν και να οριστούν οι οριακές τιμές και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. κύριος Μαρτσικέβιτς, λοιπόν, τελευταίος ομιλητής, θα μιλήσει για δύο λεπτά. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε δύο πτυχές. Καταρχάς, 3-2. 3-2 ο αγώνας της πρώτης Ολλανδίας με την Παραγουάη. Και δεύτερον, η νομοθεσία με την οποία έχουμε να κάνουμε σήμερα βελτιώνει και την ενεργειακή μας στρατηγική. Μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την, ε, τις εκπομπές ρήπων. 90% των αναγκών μας σε ενέργεια στην Πολωνία καλύπτονται από την καύση του άνθρακα. Άρα είναι βέβαιο ότι δεν έχουμε επαρκή ασφάλεια ενεργειακή στην Πολωνία. Χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος, εξαίρεση δηλαδή, έτσι ώστε να, να μετατραπεί η βιομηχανία μας και η ενεργειακή μας παραγωγή. Και για να μπορέσουμε να ε, ανεγείρουμε νέε εγκαταστάσεις, νέε βιομηχανικέ εγκαταστάσεις, εργοστάσια, σύγχρονα, με την τελευταία λέξη τη τεχνολογία, με την πιο καθαρή τεχνολογία και αποτελεσματικά. Και επίσης επιδιώκουμε και την μεγαλύτερη διαφοροποίηση καυσίμων για την βιομηχανία μας, για την ενέργειά μας. Πρέπει να προσθέσω ότι η Πολωνία θέλει να εφαρμόσει έως το 2020 το πακέτο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και να αυξήσει το ποσοστό μέσα στον ενεργειακό της μείγμα των ανανεώσιμων πηγών μέχρι το 20%. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρσινκίεβιτς. Έχουμε τέσσερις συναδέλφους που ε, συμμετέχουν στην συζήτηση με το σύστημα του ΚΑΤΣΔΙ. Για ένα λεπτό, η κυρία Ρόιτο. Ε, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι γιατί ο συμβασμό που επετεύχθη ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο αποτελεί μια λογική λύση για να προβούμε στην αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής. Στηρίζεται σε πολιτική συμφωνία η οποία επιτεύχθη επί ε, προεδρίας, ψυχικής προεδρίας όσον αφορά την παρέκκληση ε, για τις υφιστάμενες βιομηχανίες που χρειάζονται κάποιο χρόνο για να εξυγχρονιστούν. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο λαμβάνοντας υπόψη την κρίση. Ως ε, ιατρός συμφωνώ ε, για ε, σημαντική μείωση αυτών των εκπομπών. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα εφικτό. Ε, να σας πω ότι στην Δημοκρατία της Τσεχίας ήδη έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία για τη βιομηχανία και έχουμε εθνικό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών μέσα σε 10 χρόνια. Φοβάμαι ότι η έγκριση νέων προτάσεων πέραν των πλαισίων του συμβασμού θα, θα οδηγούσε σε αποτυχία την, την αδιατύπωση. Πάντω ευχαριστώ όλους όσου διαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Θέλω να υποστηρίξω τις προσπάθειες του κύριου Κράμερ, του εισηγητή, για να υλοποιήσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Από την άλλη, κατανοώ και τις ανησυχίες των κρατών μελών, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αναγνωρίζεται η δυσχερής κατάσταση ορισμένων κρατών μελών. Η παραγωγή η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής μπορεί να είναι ένα παράδεκτο κόστος ε, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, ειδικά σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα μολυσμένες. Θα πρέπει παρόλα αυτά να ε, συνεχίσουμε την άσκηση πίεσης για να εξυγχρονίσουμε τις μεθόδους παραγωγής και να έχουμε επικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, ούτως ώστε να ε, εφαρμόσουν αυτή τη φιλοσοφία και να την κάνουν έργο ε, στις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις. Κόρτινγκερ, ε, η κυρία Κόρτινγκερ έχει το λόγο. Η απλούστευση κατάρρευση της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματικότερη λειτουργία είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της οδηγίας που θέλουμε να τροποποιήσουμε τώρα για πιο αποτελεσματική πιο αποτελεσματικό περιορισμό των ρηπογόνων εκπομπών από τη βιομηχανία. Χρειάζεται κατάρριση τη γραφειοκρατία, χρειάζεται μια σαφή, κωδικοποιημένη και συμπαγή νομοθεσία, η οποία να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεσματική εφαρμογή τη για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντο μα. Και ταυτόχρονα η τήρηση των ε, νέων οδηγιών πρέπει να επαληθεύεται ότι όντω ε, εφαρμόζεται, υπάρχει. για την προστασία του, από τις κλιματικές αλλαγές, ε, την προστασία του περιβάλλοντος, ε, βαρύνοντα ρόλο έχει να διαδραματίσει και η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα και η βιομηχανία έχει ε, να συμβάλλει από πλευρά τη με τη μείωση των ρηπογόνων στην προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαρινέσκου. Κύριε Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι το συμβαστικό κείμενο είναι πολύ καλό γιατί εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ κρατών ε, μελών σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμοστική νομοθεσία. Υπάρχουν επίσης διευκολύνσεις για τις εταιρείες που δεν μπορούν, τις βιομηχανίες που δεν μπορούν να τηρήσουν τα πρότυπα μέχρι την προθεσμία. Υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει όμως να εφαρμόσουν οι πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαιρέσεις μπορούν να δοθούν για τις ε, οριακές τιμές σε περίπτωση που το κόστος ε, για τη μείωση των εκπομπών είναι πάρα πολύ υψηλό και δεν το δικαιολογούν τα ωφέλη τα περιβαλλοντικά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν όχι μόνο το, την περιβαλλοντική προστασία και εδώ διακόπτει ο πρόεδρος του ομιλητή. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε αυτό το νομοθετικό πακέτο. το οποίο θα πρέπει να έχει κάποια περιβαλλοντικά ωφέλη. Η οδηγία αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις, ε, τεχνικές. Ε, δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει ο, ο, δεν να ε, παρακολουθήσουν οι διερμηνείς, γιατί μιλάτε με τέτοια ταχύτητα που είναι αδύνατο να σας παρακολουθήσουμε. Θα πρέπει οι εγκαταστάσεις να κλείσουν ε, συχνά πολύ γρήγορα και το κόστος για τους καταναλωτές θα είναι τεράστιο. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν, λοιπόν ένα συμβιβασμός ανάμεσα στο περιβάλλον και στο κόστος για τις επιχειρήσεις. Ε, είναι καλό που θα έχουμε όρια στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με, το, με τη διαδικασία του Catch the Eye. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Ποτότσνικ για να αντιδράσει στις ε, παρεμβάσεις. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα τη προστασία του περιβάλλοντο και τη τρέβλωση του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Καταρχά, θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για τη χορήγηση των αδειών και κριτήρια για την θέση των οριακών τιμών εκπομπών. Η ευελιξία είναι δυνατή, αλλά θα πρέπει να δικαιολογείται. Η Κομισιόν πρέπει να συλλέγει πληροφορίε για τη χρήση αυτή τη ευελιξία. Οι μεγάλε πηγέ ε, ρήπανση, οι μεγάλε εγκαταστάσει καύση θα πρέπει να εφαρμόσουν τις βέλτιστες ε, διαθέσιμες τεχνικέ μέχρι το 2020 ή αλλιώς να κλείσουν μέχρι το 2023. Θα γνωρίζετε βεβαίω ότι ε, έτσι έχει η πρότασή μας. Όλα αυτά τα μέτρα, καθώς και τα μέτρα για τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, σημαίνει ότι το πακέτο αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Η Κομισιόν είναι έτοιμη για να προχωρήσουμε στη φάση της εφαρμογής. Έχω τονίσει κατά επανάληψη ότι δεν θα διστάσω για να ξεκινήσω διαδικασίες επί παραβάση αν χρειαστεί. Ελπίζω και νομίζω ότι το έχω αποδείξει ε, στο πρώτο μισό της ιτίας μου ότι η ισοτιμία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ισοτιμία απέναντι σε... και δικαιοσύνη απέναντι σε όλου. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Φυσικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και φυσικά θα πρέπει να ανταγωνιστούμε με την Κίνα και να είμαστε θέσει να ανταγωνιστούμε, αλλά όχι με τα δικά του πρότυπα για τον αέρα. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ πρόοροι θάνατοι και έχει αποδειχθεί ότι προκαλούνται από, κακές, από κακής ποιότητας αέρα. Εντάξει, να δώσουμε χρόνο στη βιομηχανία για να υπάρξουν αλλαγές, να ενσωματώσουν τις αλλαγές, αλλά θα πρέπει να δούμε και τη θετική πλευρά της όλης προσπάθειας, ότι κερδίζουμε και τεχνολογικά, τεχνολογικά, τεχνολογική, σε τεχνολογική προσπάθεια, σε τεχνολογική πρόοδο. Ε, ούτως ή άλλως η αρχική πρόταση βασίστηκε σε μια μελέτη αντικτύπου που έγινε μέσα σε δύο χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη ε, και συμμετείχαν πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί των κρατών μελών. Η έννοια των βέλτιστων τεχνικών είναι σημαντική. Επίσης, έχουμε πολλές συμπληρωματικές πολιτικές για να υποστηρίξουμε τη βιομηχανία. Ε, σχέδια δράσης για το περιβάλλον, προγράμματα για την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, ε, διαρθωτικές επιδοτήσεις κτλ. Επομένως, ε, αν έχουμε καλύτερο περιβάλλον, περισσότερες ε, θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μείωση του κόστους, αυστηρότερους κανόνες, περισσότερη ευελιξία, και εξισορρόπηση των συμφερόντων. Όλα αυτά είναι στοιχεία του συμβιβασμού. Το θέμα είναι ότι κινούμαστε και κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Ε, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ε, πιο υγιές περιβάλλον, ε, περισσότερη δικαιοσύνη για τη βιομηχανία, περισσότερα κίνητρα για την καινοτομία. Και νομίζω ότι τελικά η πρόταση που είναι επιτάπητος ε, η οποία, την οποία εκπώνησε ο εισηγητής είναι θαυμάσια και αξίζει τη υποστηρίξή σας. Η Κομισιόν τουλάχιστον θα την υποστηρίξει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ τώρα, ο εισηγητής έχει δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατέστησα σαφές όσο συζητούσαμε ότι ε, θα είναι Ευρωπαίος ο πρωταθλητής ε, ποδοσφαίρου εφέτος. Δεύτερον, λάβαμε ε, συγχαρητήρια από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το περιμέναμε. Και τρίτον, φαίνεται ότι και οι πράσινοι έχουν βρει τη θέση στον κόσμο γιατί είναι πιο σημαντικό το ποδόσφαιρο από την προστασία του περιβάλλοντο. Πρέπει και αυτό να το διαπιστώσουμε με ικανοποίηση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη χρήσιμη συζήτηση. Για τη συζήτηση όμω τώρα πραγματοποιήθηκε, θα ήθελα να πω τα εξή. Πρώτον, αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες και επιφυλάξεις ε, των συναδέλφων από την Ανατολική Ευρώπη με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ανατολικοευρωπαίος είμαι κι εγώ, από την Ανατολική Γερμανία. Καταλαβαίνω ότι κάθε βήμα που ολοκλήρωσαν σε δεκαετίες μέσα τα παλαιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς καλείστε να το πραγματοποιήσετε πολύ πιο γρήγορα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να προσαρμοστείτε σε νέες συνθήκες τόσο γρήγορα. Ναι, αλλά η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν τα κράτη αυτά νομίζω καλύπτεται ικανοποιητικά από τον συμβιβασμό. Και δεύτερον, δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν οι βέλτιστες ε, διαθέσιμε τεχνικές να αποτελούν κίνδυνο για τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητά μα έναντι τη Κίνα ιδιαίτερω. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδου επιχειρήματα. Είμαστε σε θέση να ε, αντέξουμε στα φθηνότερα ούτως ή άλλως προϊόντα των κινέζικων ε, βιομηχανιών ή των βιομηχανιών των άλλων των δουλικών κρατών της Ασίας μόνο και μόνο επειδή έχουμε καλύτερα προϊόντα και γιατί διαφυλάσσουμε υψηλά επίπεδα ε, ποιότητας του περιβάλλοντος και κανέναν άλλο λόγο. Έχουμε επαρκείς λοιπόν μεταβατικές περιόδους. Δεν ζητούμε μέσα σε μια εβδομάδα να ε, προσαρμοστούμε στι νέε συνθήκε και προδιαγραφέ. Αλλά το να λέει κανεί ότι για λόγους ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να εγκριθούν αυτέ οι διατάξει. δεν νομίζω ότι είναι καν λογικό σε όρου ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ και συγχαρητήρια για την πολύ καλή σα δουλειά. Η, συζήτηση η, ολοκληρώ... η συζήτηση ολοκληρώθηκε, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι πλέον και το τελευταίο τέτοια ώρα.